Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης, την εκλογή δηλαδή αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω λάβει τα εξής ονόματα υποψηφίων. Ρομπέρτα Αντζελίλη. Μπέλ. Καμίνσκι Μίχαου Τόμας. Κοχ Μέριν Σιλβάνα. Κράτσα Τσαγκαροπόλου. Ρόντι. Λαμπρινίδης Σταύρος. Μακμίλαν Σκοτ Ιντουόρτ. Μαρτίνες Μαρτίνες Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rodberend Dagmar, Rouczek Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów Έχουμε περισσότερους δηλαδή από 14 υποψηφίους ενώ είναι 14 οι αντιπρόεδροι οπότε θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία στον πρώτο γύρο της ε, ψηφοφορίας οι δε καταμετρητές των ψήφων θα είναι ακριβώς οι ίδιοι που ήταν και για την εκλογή του Προέδρου, οπότε σας παρακαλώ να μετακινηθείτε στις κάλπες και να θυμάστε ότι θα ψηφίσετε τελευταίοι. Επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού, επειδή έχουμε περισσότερους υποψηφίους αποθέσεις, θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία. Διαβάζω το ε, σχετικό άρθρο. Όλοι χρησιμοποιούν μόνο μία κάρτα και επιλέγουν το άτομο το οποίο θέλουν να ε, ψηφίσουν. Σας παρακαλώ καθίστε γιατί διαβάζω άρθρα από τον ε, κανονισμό και το τι πρέπει να γίνει τα επόμενα 20 λεπτά. Στον, ε, στον πρώτο γύρο έχουμε 14 θέσεις. Όσοι υποψήφοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων θα